Euh, Ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις, για τις παρεμβάσεις σας λοιπόν. Ε, τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε ένα άλλο θέμα πιο τεχνικό αυτή τη φορά για ένα θέμα επικουρικότητας. Για να αρχίσουμε τη συζήτηση θα δώσω το λόγο καταρχάς στον Μάριο Μπορκέτσιο για τέσσερα λεπτά. la posizione del gruppo che io rappresento, FD, è molto chiara. Si chiede con questa interrogazione orale alla Commissione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 να έρθω στην ουσία αυτής της ε, απόφασης ε, που δεν ε, μπορεί να θεωρηθεί πράξη δημοκρατίας και ελευθερίας όπως υποστηρίζουν περισσότερο. Είναι πράξη αστυνόμευσης της σκέψης, μια αντιδημοκρατική πράξη. Αν μέσα στο, στον τοίχο μιας σχολικής αίθουσας υπάρχει ένα σταυρός και αυτός αφαιρεθεί, αυτό δεν είναι ε, ένας τείχος λαϊκός, είναι ένα τείχος άδειος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα από τα πολλά δείγματα ε, πνευματικής αυτοκτονίας της Δύσης. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου ε, θεωρεί ότι υπάρχει ένα είδος ε, θρησκευτικής ελευθερίας που αν φτάσει στα όρια της θα έπρεπε να υποχρεώσει κάθε πολίτη να ζει σε ένα περιβάλλον σύμφωνο με το πιστεύω τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι η θρησκευτική ελευθερία. Ε, εδώ, αντίθετα, έχουμε ένα αρνητικό δικαίωμα. Ένα ε, δικαίωμα να ε, ελεγχόμαστε όσον αφορά τη θρησκευτική μας συμπεριφορά. Ε, όταν μιλάμε για το θρησκευτικό αίσθημα, μιλάμε για κάτι όχι ε, το, τόσο συγκεκριμένο. αλλά ο Σταυρός ε, δεν είναι συμβολοποίηση μόνο στον πολιτισμό μας. Είναι κάτι πιο σημαντικό, είναι κάτι το παγκόσμιο, ε, το καθολικό. Ο συμβολισμός του Σταυρού έχει μία εμβέλεια ε, παγκόσμιου μηνύματος, μηνύματος αδελφοσύνης, μηνύματος ειρήνης, όπως μας έχουν διδάξει οι μεγάλοι σοφοί. Από την άποψη αυτή λοιπόν είναι σαφέστατη η αξία του Σταυρού. Αλλά μιλώντας για αυτή την απόφαση έχουμε να κάνουμε με στάσεις που οδηγούν προς μια ομοιομορφία της σκέψης. Είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το πραγματικό πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πραγματικά απίστευτο που συμβαίνει. Ε, σαν ε, το αίτημα ήταν να αποσπαστούν οι λαοί μας από κάθε αξία, κάθε σύμβολο που μας σβρώχνει προς την πνευματικότητα πέρα των ιστορικών ε, γεγονότων, ε, του ιστορικού δεδομένου ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη θρησκεία. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο σύμβολο, επαναλαμβάνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, θα πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των λαών να χρησιμοποιούν τα σύμβολα, ε, ξεκινώντας από το Σταυρό. Θα πρέπει να έχει το κουράγιο η Ευρώπη για αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα να υιοθετήσει μια προοπτική μεταιστορική, να ε, αναλάβει ε, το ρόλο της σαν πνευματικό κέντρο να εξασφαλίσει στους ευρωπαϊκούς λαούς ε, για τους ευρωπαϊκούς το δικαίωμα να διατηρήσουν τα σύμβολά τους και την πίστη τους ε, μέσα στην νομικο δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας και όλο το ζήτημα στρέφεται γύρω από αυτό το θεμελιώδες ζήτημα της αρχής της επικουρικότητας. Ολοκληρώνω. Το θέμα αυτό μας επιτρέπει να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε το πολύ κεντρικό ζήτημα που είναι τι είναι για την Ευρώπη η έννοια της, της θρησκευτική ελευθερίας, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου καταπάτησε την ελευθερία του θρησκευτικού αισθήματο. Πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα ε, να, παραμείνουν, ε, να παραμείνει ο σταυρό στι σχολικέ αίθουσε, διότι αυτή είναι η παράδοσή μα, αυτέ είναι οι ρίζε μα. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρο. Νομίζω ότι καταλάβαμε το νόημα τη παρέμβασή σα. Για δύο λεπτά ο κύριο Αντώνιο Καντσιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, στις 3 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, δέχτηκε μια προσφυγή ε, μιας ε, Ιταλοφιλανδέζας με σκοπό να αφαιρεθεί ο Σταυρός από τις σχολικές αίθουσες. Παρόμοια συμβάντα έγιναν στο παρελθόν στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία αλλά και στην Ιταλία οπότε το 88 ένα δημοτικό συμβούλιο ε, αφαίρεσε ε, τον ε, κατέργησε το Σταυρό. Το Συμβούλιο Επικρατείας το 2006 στην Ιταλία διευκρίνησε ότι η αρχή ε, του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη την πολιτιστική ταυτότητα και τον πολιτισμό ενός λαού. Με την ερώτησή μας θελήσαμε να εντοπίσουμε ακριβώς τον πιο λαϊκό χαρακτήρα αυτού του ζητήματος και να θέσουμε και μια πρόκληση ότι το επόμενο βήμα ε, θα μπορούσε να είναι όλα τα σύμβολα ε, καθολικής έμπνευσης που είναι κοινά στα κράτη-μέλη καθώς επίσης και οι πολιτικές και καλλιτεχνικές εκφράσεις που υπάρχουν σε αυτονία στις χώρες μας να ε, απαγορευτούν ακόμα και οι σημαίες ε, ε, των ευρωπαϊκών κρατών. Ε, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσπαθεί να επιβάλλει ένα μοντέλο λαϊκότητας που δεν μπορεί να είναι το δικό μας. Μακριά από την αρχή της επικουρικότητας αυτό είναι ο, ο κενός τείχος που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος. Αφιζητείται και διακυβεύεται η ίδια μας η ταυτότητα, οι αρχές μας, ε, της ειρήνης, της αγάπης, της κοινωνικής ειρήνης, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Η απόφαση αυτή είναι μια ε, ενέργεια κατά της ε, ελευθερίας και των δικαιωμάτων. Ε, η, η έκθεση των πολιστικών και θρησκευτικών συμβόλων μέσω των οποίων ο λαός αναγνωρίζει την ε, ελευθερία της ε, σκέψης του. Είναι ιερά και απαραβίαστα και έτσι πρέπει να τα υπερασπιστούν τα ίδια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που βασίζονται ε, στις δημοκρατικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μάουρο Μάριο. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ε, προηγουμένως ο κύριος Επίτροπος. Πολύ ευχαρίστω να ακούσω τον κύριο Μάουρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάρει το λόγο μετά από μένα. Είμαι υποχρεωμένο ε, να ακολουθήσω ορισμένου κανόνε δικαίου. Η Κομισιόν ασφαλώ υποστηρίζει την ελευθερία σκέψη, την ελευθερία συνείδηση και θρησκευτική ελευθερία, όπω προβλέπεται το άρθρο 9 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 ε, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια όμω είναι ότι η Κομισιόν μπορεί να δράσει μόνο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, του κοινοτικού δικαίου. Και στο, το κοινοτικό δίκαιο ε, προβλέπει ότι ε, τα θέματα τα σχετικά με τα σύμβολα στα δημόσια κτίρια αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η αρχή της ε, κορικότητα εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι αλήθεια ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται στην εφαρμογή της εκτέλεσης μιας απόφασης του ΔΕΚ ε, από τις ε, εθνικές αρχές οι οποίες πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι αλήθεια ότι η εκτέλεση των αποφάσεων του ε, είναι ε, αρμόδια της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να σέβονται τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 43, οι Ιταλικές Αρχές έχουν ένα μήνα ε, προκειμένου να ε, ζητήσουν να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, η Ιταλία ε, ζήτησε να παραπευθεί η υπόθεση, έκανε έφεση δηλαδή κατά πάση. Εμείς από την άλλη πλευρά μπορούμε να εφαρμόσουμε, μάλλον περιοριζόμαστε από την εσωτερική ενωμητάξη των κρατών μελών. Εγώ δεν μπορώ να υποκαταστήσω ούτε το Συμβούλιο ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Που πήρε μια απόφαση η οποία κατανοώ ότι μπορεί να δημιουργεί κάποια προβλήματα ή κάποιες ανησυχίες. Αυτά σας τα λέω ειλικρινά. Τι άλλο να πω. Θα ακούσω και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Φαλώς με προσοχή. Ωραία, ο λόγος στον κύριο Μαύρο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την σαφήνεια της ε, κρίσης που εξέφρασε και που παραπέμπει το θέμα αυτό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά είμαι πεπισμένος, όπως λίγοι άλλοι, σχετικά με την ανάγκη του λαϊκού χαρακτήρα των θεσμών μας. Και είμαι επίσης πεπισμένος ότι η θρησκεία δεν είναι η λύση κανενός πολιτικού προβλήματος. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να βρεθεί η λύση των πολιτικών προβλημάτων ε, μέσα από τον πόλεμο ε, ενάντια στη θρησκεία. Θα εκφράσω την σκέψη μου μέσω ενός παραδόξου. Τι θα συνέβαινε αν εφαρμόζαμε την απόφαση του Στρασβούργου. Δηλαδή αν εφαρμόζαμε αυτή τη λογική που επιβάλλει την κατάργηση του Σταυρού από τις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας παράλληλα για, σε όλους τους τόπους όπου υπάρχει ε, δημόσια ε, παρουσία του Σταυρού. Τι θα κάνουμε με τη σημαία της ε, Σουηδίας, με τη σημαία της Φιλανδίας που σας δείχνω εδώ. Τι θα κάνουμε με τη σημαία της Σλοβακίας, τη σημαία της Μάλτας, της Δανίας της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχει τρεις σταυρούς μάλιστα. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ο λόγος που υπάρχουν αυτοί οι σταυροί σε αυτές τις σημαίες δεν είναι διαφορετικός από το λόγο για τον οποίο υπάρχει ο σταυρός στα σχολεία της Ιταλίας. Δεν είναι θρησκευτικός ο λόγος, είναι ο λόγος πολιτισμού και παραδόσεων. Ας αφήσουμε λοιπόν να είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία θα κρίνουν κατά περίπτωση την ε, ορθότητα των λύσεων που να ταιριάζουν στο λαό της κάθε χώρας με σεβασμό της θρησκευτική ελευθερίας και με σεβασμό στο, προς το λαϊκό χαρακτήρα των θεσμών. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Και το ζητάμε αυτό γιατί πριν, πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρχει σεβασμός για την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου πάνω και από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Ο λόγος του κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ. Ως νομικός και ως μέλος του Κοινοβουλίου συμμερίζομαι με πολλούς από τους πολίτες μας ε, την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ενώπιον ε, μιας ε, συζήτησης άστοχης. Ας διευκρινίσουμε σημαντικά πράγματα. Πρώτον, Μιλούμε για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται για όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα αυτόνομο όργανο ε, σε ένα πλαίσιο ομόκεντρων κύκλων, αλλά όχι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, μιλούμε για ε, ένα, μια δικαστική απόφαση και καμία απόφαση του δικού μας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί, δεν μπορεί να αλλάξει, να τροποποιήσει, να καταργήσει αυτην την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τρίτον, αυτή η απόφαση ε, σέβεται την θρησκευτική ελευθερία και την κορονίδα της, ε, την το θρησκευτικό πλουραλισμό, τη θρησκευτική πολυφωνία. Σέβεται το συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών, ε, μάλλον η, ελευθερία αυτή ε, γίνεται σεβαστή από το, το Σύνταγμα των Κρατών Μελών και από ε, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, η απόφαση αυτή δεν αρνείται τη θρησκευτική ελευθερία και ε, μάλιστα ελήφθη αυτή η απόφαση ομόφωνα από ένα δικαστήριο ψηλού κύρους που έχει προσπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα τα τελευταία 60 χρόνια. Τέλος, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι καμία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων δεν ε, ε, οδηγεί στην τροποποίηση οποιασδήποτε νομοθεσίας κράτους μέλους διότι αναγνωρίζει μόνον ε, βλάβη ε, η προσβολή των δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το κράτος μέλος μετά μπορεί να αλλάξει αν θέλει την νομοθεσία του εμπνεόμενο από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων αλλά καμία απόφαση δεν απαιτεί από τα κράτη-μέλη να αλλάξουν την νομοθεσία τους κανένα κράτος που έχει υπογράψει τη ε, Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν υποχρεούται να αλλάξει την νομοθεσία του κατόπιν αποφάσεως του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνεπώς ούτε η Ιταλία ούτε καμία άλλη χώρα θα πρέπει να πάρει μέτρο γενικού χαρακτήρα. Τέλος, μιλώντας για την επικουρικότητα. Η επικουρικότητα αποτελεί ένα κανόνα δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που όμως δεν εφαρμόζεται επουδενή σε αυτήν την περίπτωση διότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να επικαλούμεθα ένα κανόνα του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κοινοτικού δικαίου, ε, για να αμφισβητήσουμε ε, μία απόφαση η οποία δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού, του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, η συζήτηση αυτή είναι άκερη, είναι άστοχη και ε, δεν υπάρχει κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο λίγο λόγο στην κυρία Σόφια Ιντβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο παραπλανητικό τίτλο τη σημερινή συζήτηση περιλαμβάνει την λέξη επικουρικότητα. Η επικουρικότητα, όπω την καταλαβαίνω εγώ, είναι να λαμβάνονται αποφάσει στο πιο εγγύς επίπεδο προ τον πολίτη. Και το επίπεδο αυτό, συνάδελφοι, είναι ο πολίτης, ο κάθε πολίτης. Αυτό που λέμε στο ψήφισμα αυτό είναι ότι το δικαίωμα του εθνικού κράτους υπερισχύει του δικαιώματος του πολίτη και είναι δική μας δουλειά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο να προστατεύουμε τα δικαιώματα του πολίτη, όχι τα δικαιώματα του κράτους. Κατά δεύτερον, αν όπως ισχυρίζεστε θεωρήσουμε ότι δεν πρόκειται για θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταλάβω γιατί περιλαμβάνεται τότε στα κριτήρια τη Κοπενχάγης, γιατί ζητάμε από τις υποψήφιες χώρες να σεβαστούν την διάκριση εκκλησίας και ε, κράτους, όταν δεν μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό από τα κράτη-μέλη μας. Και αν λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο να μιλά για τέτοια θέματα, αναρωτιέμαι γιατί μπορούμε να συζητάμε θέματα όπως το σχήμα των αγκουριών και όχι θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μας. Επειδή η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η απόφαση του Δικαστηρίου Δύο εβδομάδες τώρα μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά και την ε, συμπερίληψη του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα έπρεπε να αρνηθούμε να... Πώς μπορούμε να αρνούμαστε την ε, ε, αρμοδιότητα του δικαστηρίου του Στρασβούργου και κατά δεύτερον οι πολιτικοί δεν έχουν... δεν μπορούν να μειγνύονται τις δικαστικές αποφάσεις σας, κάνουν οι δικαστές τη δουλειά τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν έχουμε δικαίωμα να εμπλεχτούμε. Εγώ από τους φιλελευθέρους θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι για όλους τους πολίτες και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα συνείδησης, θρησκείας και αν θέλετε και έχει δικαίωμα να μην έχει θρησκεία. Τα κράτη είναι αυτά όχι τα δικαστήρια τα οποία θα πρέπει να διασφαλίσουν ένα περιβάλλον όπου θα μπορούν ελεύθερα να ζουν οι πολίτες κατά τη συνείδησή τους. Θα πρέπει να προστατεύονται από τα κράτη αυτά. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση τη στιγμή που αισθάνονται την ανάγκη να, προς, να πάνε στα δικαστήρια. Συνάδελφοι, προτείνω να, να απορρίψετε αυτό το ψήφισμα. Ο λόγος στον κύριο και για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεδομένων των ιστορικών γεγονότων, βάσει των οποίων οι ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Αντενάουερ, Μονέ, Σούμαν, ε, ήταν χριστιανοδημοκράτε, όλοι του βασίστηκαν στα χριστιανικά σύμβολα και αξίε. Οι, σημαίε που, οι που βρίσκονται πίσω από την κυρία Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η σημαία της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, αναφέρεται στα 12 αστέρια πάνω από το κεφάλι της Παρθένου Μαρίας. Η απόφαση αυτή είναι σκανδαλώδης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Και απέναντι στην απόφαση αυτή πρέπει να πούμε ότι κανένας δικαστής που ορίστηκε από τους πολιτικούς δεν μπορεί να απαιτήσει την άρνηση του Σταυρού. Υιοθετώντα την ε, απόφαση αυτή, απαρνούμαστε τις χριστιανικές αξίες. Κύριε Επίτροπε, δεν πιστεύετε ε, ότι πρόκειται για μια ενέργεια κατά των χριστιανικών αξιών και ότι αυτό θα οδηγήσει την Ευρώπη στην καταστροφή δεν θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με την αξία, ε, τη σημασία των ε, χριστιανικών αξιών ε, στην Ευρώπη. Ο κύριος Βέμπερ. Να σας ευχαριστήσω για τη διεξάγωγη τη συζήτηση αυτή. Ο συνάδελφος Λόπες είπε ότι ως νομικός δεν είμαστε αρμόδιοι. Εγώ δεν μιλάω ως νομικός, μιλάω ως πολιτικός. Εκατομμύρια ε, κόσμος πλήττεται στην Ευρώπη από την απόφαση αυτή και πιστεύω ότι είναι καλό να το συζητήσουμε. Δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω. Η σχέση μεταξύ Εκκλησίας και κράτους στην Ευρώπη πάντα ήταν αμφιλεγούμενη και οδήγησε σε αιματηρές συγκρούσεις. Είναι σωστό λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατάφερε να χωριστεί το κράτος και η Εκκλησία ορθό και σωστό. Στην Ευρώπη, ε, κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά διαφορετικά μοντέλα. Στην ε, Γαλλία έχουμε κοσμικό χαρακτήρα, στην Μεγάλη Βρετανία η Βασίλισσα είναι η ύπατη εκπρόσωπος της Εκκλησίας και υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα για τη σχέση αυτή μεταξύ κράτους και Εκκλησίας και νομίζω ότι είναι σωστό να εφαρμόσετε εδώ η επικουρικότητα. Κάθε χώρα να ακολουθεί το δικό της δρόμο και θα ήθελα να πάω και ένα βήμα παραπέρα, όχι να μιλήσουμε μόνο για το θέμα της επικούρικότητα, αλλά για το βασικό θέμα για τα θέματα αλληλεγγύης, ελευθερίας, επικουρικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς βάση στο χριστιανισμό δεν νοούνται αυτές οι αρχές. Γιατί υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν ε, με τον τρόπο αυτό οι αρχές αυτής στον αραβικό κόσμο, στην Κίνα. Γιατί βασίζονται, έχουν τις ρίζες τους στη δική μας θρησκεία. Είμαστε περήφανοι για την ε, ανεξιθρησκεία που επικρατεί στην Ευρώπη, αλλά κυρίες και κύριοι, η ανεξιθρησκεία εκφράζεται με το να επιλέγει κανείς να είναι άθεος, για παράδειγμα. Αυτό είναι απόλυτα νόμιμο, αλλά υπάρχει και το δικαίωμα να έχει κανείς πίστη στη δική μου περιφέρεια με παραπάνω από ένα εκατομμύριο ψήφοφο πολίτες πάνω από 80% του πληθυσμού είναι καθολικοί. Όπως αποδεχόμαστε για το δικαίωμα του άθεου να είναι άθεος, έτσι αποδέχεται και ο άθεος το δικαίωμα του καθολικού να είναι καθολικός και σε αυτό σου και η αποδοχή των χριστιανικών συμβόλων. Και αυτό είναι νόμιμο και δικαιολογείται από το δικαίωμα της ε, για όσους δηλαδή εκπροσωπούν τη χριστιανική πίστη. Ευχαριστούμε κύριε Βέμπερ. Και τώρα η κυρία Σενιζίν. Pani Przewodnicząca, koleżanki. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Αθλητικών Δικαιωμάτων του Στρασβούργου ε, πολύ ορθά είπε ότι οι σταυροί στα σχολεία παραβιάζουν την θρησκευτική ελευθερία των μαθητών και των γονέων τους. Οι δικαστές ε, ε, ανέφεραν ότι η παρουσία αυτών των σταυρών αντιβαίνει με, την, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ε, οι πολιτικοί της ε, δεξιάς κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ζητούν εξηγήσει από την Κομισιόν, ε, αλλά δεν είναι αυτός ο ορθός δρόμος. Τα ευρωπαϊκά όργανα δεν έχουν να κάνουν τίποτα ε, σε σχέση με αυτή την απόφαση. Το δικαστήριο αυτό αποτελεί όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση σχετική με τους σταυρούς δεν αντιβαίνει με την αρχή της επικουρικότητας. Αντιθέτως, επιτρέπει να ε, εφαρμοστεί το δίκαιο στις ε, χώρες οι οποίες ε, προβλέπουν το χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Η απόφαση αυτή λοιπόν θα βοηθήσει στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών έναντι της ε, ε, ε, αυξανόμενης τρισκοληψίας που χαρακτηρίζει ορισμένες κοινωνίες. Η απόφαση αυτή δεν πλήττει την κοινωνική ταυτότητα ή την εθνική ταυτότητα των οποιασδήποτε χώρας. Γιατί μιλούμε μόνον για τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία. Κανένας δεν ζήτησε, για παράδειγμα, να καταργηθεί ο Σταυρός από τις σημαίες. Προφανώς όχι. Κανένας δεν επιτίθεται στην Εκκλησία. Απλώς υπερισπιζόμαστε τα δικαιώματα των πολιτών. Η κατάσταση ενίσχυσης ε, του κλήρου και των ε, και τη εκδήλωση των θρησκευτικών δικαιωμάτων πλήττει τα δικαιώματα άλλων σε χώρε όπω η δική μου Πολωνία. Οποιαδήποτε απόφαση αμφισβήτηση θα μα γελιοποιήσει. Ευχαριστώ. Ο λόγο του κ. Καζίνη για δύο λεπτά. Η απόφαση του δικαστηρίου ε, ενόχλησε όλους αυτούς που στο Σταυρό εδώ και αιώνες βλέπουν ένα σύμβολο ε, ελπίδας, ανακούφισης από το φόβο και από ε, τα βάσανα. Εμείς ζητήσαμε να γίνει αυτή η συζήτηση για να είναι, γίνει σαφής η λογική. Τι πρέπει να βγάλουμε, να αφαιρέσουμε τους σταυρούς που βρίσκονται ε, και δεσπόζουν στις πόλεις μας πάνω στις εκκλησίες και στα μέγαρα. όλα αυτά προκαλούν ένα προβληματισμό πάρα πολύ σημαντικό και από την άποψη των δικαιωμάτων των πολιτών και από την πολιτική άποψη. Τα δικαιώματα ε, είναι ατομικά δικαιώματα ε, ή δικαιώματα ενός λαού που θέλει να εκφράσει τη θρησκευτικότητά του. Δεν μετράει σε τίποτα η ιστορία, ο πολιτισμός, η τέχνη που επί αιώνες έχουν ε, σημαδέψει έναν λαό. Και φυσικά υπάρχει θέμα επικουρικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ε, υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αξίες που θεωρούνται παγκόσμιες, βέβαια, καθολικής ε, ισχύω, αλλά μπορεί να υπάρχουν και συγκρούσεις ανάμεσα στα δικαιώματα. Γιατί να αρθεί το δικαίωμα των κρατών μελών να λύνουν τέτοια προβλήματα, ανάλογα με τις ευαισθησίες και τις παραδόσεις του λαού τους. Το θέμα λοιπόν ξεπερνάει το ζήτημα του Σταυρού απλώς. Υπάρχει ε, αναγνώριση ε, των αρμοδιοτήτων των κρατών. Όπως θα για το θέμα της ε, ε και της ευθανασίας. Όμως, η συνθήκη της Λισαβόνας μας υποχρεώνει να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόσφαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο για αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό ε, εκφράζει ε, ένα μικρό ρυθμό ε, ανθρώπων και αυτό σίγουρα παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι τελικά η απόφαση αυτή ενάντια στα δικαιώματα και στην ελευθερία. Ευχαριστώ κύριε Καζίνη. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Καταρχήν ο λόγος του κύριο Μικολάζικ. Για ένα λεπτό. Dejiny Európy, jednotlivých štátov a teda Európskej únie sú, Είτε μας αρέσει είτε όχι, ε, είμαστε πολύ κοντά στον χριστιανισμό και σε πολλά συντάγματα αναφέρεται η χριστιανική παράδοση και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αρχικά. Μεταξύ άλλων υπήρχε αναφορά στο κληροδότημα του χριστιανισμού σε ό,τι αφορά τις καθολικές αξίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα τα θεμελιώδη δικαιώματα υπερασπίζονται από τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά πηγάζουν κυρίως από τις συνταγματικές παραδόσεις οι οποίες αποτέλεσαν καρπό αιώνων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί τις παραδόσεις αυτές και τις αξίες αυτές και να μην επιτρέψει να τιμωρηθούν τα κράτη-μέλη που προασπίζονται των δικαιωμάτων τους αυτούς και σέβονται μεταξύ άλλων και τα χριστιανικά σύμβολα και τη χριστιανική κληρονομιά τους. Θα ήθελα να πω τέλος ότι ούτε στις διατάξεις της σύμβασης ούτε στο χάρτη αναφέρονται τέτοια δικαιώματα señora presidenta. Καταρχήν να αναφέρω κάποιες ε, λέξεις που δεν είναι δικές μου. Ε, ο Σταυρός ε, μεταδίδει θετικές αρχές, αποτελεί τίμα της ιστορίας μας, αποτελεί ιστορία της κοινωνίας που χρονείται εδώ και χίλια χρόνια. Ε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτές τις αρχές που μας δημιούργησαν. Η δημοκρατία ε, η λειτουργεί μέσω του σεβασμού και της ελευθερίας, διευκολύνοντας την ε, άσκηση των δικαιωμάτων, όχι μέσμων. Η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να γίνει σεβαστή και να αναγνωρίζεται από όλα τα όργανα και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. η δυνατότητα των κρατών μελών να επιδεικνύουν θρησκευτικά σύμβολα στα δημόσια κτίρια όταν αυτά ε, αντικατοπτρίζουν τις ε, αρχές δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Η θρησκεία είναι ο πυλώνας στον οποίο βασίζεται η ελευθερία μας και η δημοκρατία μας. Αν αμφισβητηθεί αυτή η ελευθερία, αμφισβητείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Πανικολάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ και εγώ πως το δικαστήριο κρίνει λάθος με το να εξισώνει την παραμονή του εσταυρωμένου στις σχολικές αίθουσες με την ασέβεια προς τη θρησκευτική πίστη των άλλων. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι περισσότερο κοινωνικό παρά νομικό και είναι δεδομένο ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στην αρχή της επικουρικότητας. Η παρουσία θρησκευτικών συμβόλων δεν συνιστά ένδειξη θρησκευτικής διάκρισης ή καταναγκασμού. Πηγάζει από την παράδοση και την ιστορία της κάθε χώρας συχνά και από το σύνταγμα δε αυτής όπως συμβαίνει στη δική μου χώρα την ελλάδα. στην ελλάδα έχουμε στις σχολικές αίθουσες θρησκευτικές εικόνες όχι για να επιβάλλουμε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία στους μαθητές αλλά γιατί αποτελεί στοιχείο της παράδοσής μας άμεσα συνδεδεμένο με τις αξίες και τις δομές της κοινωνίας μας άμεσα συνδεδεμένο με τις διώξεις και τη θρησκευτική καταπίεση επί τέσσερις αιώνες από την οθωμανική αυτοκρατορία. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζεμπόσκα. Αγαπητέ Επίτροπε, συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Σήμερα, στο τέλος της χρονιάς και παραμονή Χριστουγέννων, 60 χρόνια μετά από τις, την ίδρυση της Ένωσης, ακόμα συζητάμε ένα πυλώνα της ε, Ένωση, στην αρχή της επικουρικότητας. Κατά δεύτερον, να πω ότι το θέμα είναι μία απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου σε ό,τι αφορά την παραβίαση της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης σε ό,τι αφορά την παρουσία του Σταυρού στα σχολεία στην Ιταλία. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλές ε, χώρες και η σλοβακική κυβέρνηση πριν από δύο χρόνια, πριν από δύο εβδομάδες ε, υιοθέτησε ένα ψήφισμα το οποίο αντίκειται στην ε, ευρωπαϊκή μας παράδοση και τρίτον θα ήθελα να πω ότι διαβάζοντας το ψήφισμα δεν, ενδια... δεν αισθάνομαι ιδιαίτερα καλά και λυπάμαι που δεν μπορέσουμε να εντάξουμε αυτά τα θέματα που συνδέονται με την ε, σύνθηκη της Λισαβόνας στο ψήφισμα. Ευχαριστώ. Αν ήταν ε, να εξετάσουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε τρεις και ο κούκος αυτή τη στιγμή εδώ για να μιλήσουμε για το θέμα του Σταυρού. Αν σκεφτούμε ότι για να μιλήσουμε για το Σταυρό πρέπει να επικαλεστούμε την έννοια της επικουρικότητας, δεν μπορούμε παρά να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι Βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη που ντρέπεται για την ιστορική της ε, παράδοση, για την, για την ε, ιστορική πραγματικότητα του ιουδαισμού για την ε, παράδοση μας που είναι, όπως είπε ο Γκέτε, η πραγματική κοινή γλώσσα της Ευρώπης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες που μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να κρατάει ενωμένη την Ευρώπη παρά μόνο ο χριστιανισμός. Τίποτα περισσότερο από τον χριστιανισμό. Ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο Παρό. Γιατί μετά από αυτό το δημοψήφισμα που έγινε στην Ελβετία ε, και τάχτηκε κατά του, υπέρ του όχι ε, για τους μηναέδες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισλαμική Διάσκεψη, όλοι κινητοποιήθηκαν για να καταδικάσουν αυτό το δημοψήφισμα, παρόλο που η Ελβετία δεν αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν σήμερα, ε, κατόπιν όλων αυτών, υιοθετείται μία ουδέτερη στάση για ένα θέμα που αφορά την ε, ταυτότητά μας, τις ρίζες μας, την ίδια την ψυχή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσοι είναι προτεστάντες και δεν ε, λατρεύουν το Σταυρό, εξ ονόματος λοιπόν αυτών θα ήθελα να πω το εξής, ότι προέρχομαι από μια περιφέρεια όπου το 99% των πολιτών είναι καθολικοί. Και τα παιδιά μου πάνε στο σχολείο μαζί με άλλα καθολικά Παιδιά, δεν μας ενοχλεί ο Σταυρός. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε την εξής διάκριση μεταξύ των διαφόρων συμβόλων. Δεν με ενοχλεί εμένα ο Σταυρός, ενώ άλλοι μπορεί να αισθάνεται ότι τους ενοχλεί. Στις χώρες όπου αναρτείται ο Σταυρός στις σχολικές τάξεις επειδή αυτό αποτελεί τμήμα της παράδοσης, επειδή πρόκειται για σχολεία της ε, Εκκλησίας, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συζητάμε όμως τέτοια θέματα. Θα πρέπει να συζητάμε το πώς θα βγούμε από την οικονομική κρίση, πώς θα επιλύσουμε προβλήματα σοβαρά. Γιατί α, προέβαλαν τέτοιες ενστάσεις, τέτοια παράπονα αυτοί που τα προέβαλαν στην Ιταλία, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι εμένα δεν με ενοχλεί ο Σταυρός και θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιοι όροι προκειμένου να μην ενοχλούνται οι πολίτες. Τελειώνουμε τη διαδικασία του καθιστέα με, την, με την κυρία Ντότς. In recent years we... Πρόσφατα, Έχουμε δει μια εκστρατεία καταπίεση ε, της, ε, των σκεπτικών ευθεριών. Η Λίνια Λαντέλ σήμερα, ε, πρόσφατα, έχασε την υπόθεσή της στο Ανατοδικαστήριο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου διότι η νομοθεσία δεν προστατεύει τους χριστιανούς. Η γυναίκα αυτή θα χάσει τη θέση της. Ε, ε, πριν από... Ε, μάλλον η Κομισιόν σε μια αιτιολογημένη γνώμη της ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο να περιορίσει τους, τις εγγυήσεις της σκεφτικής ελευθερίας στην νομοθεσία του κρίμα, ντροπή για την Κομισιόν. Η Κομισιόν θα πρέπει να γνωρίσει ότι οι άνθρωποι ε, έχουν το δικαίωμα να έχουν μια πίστη και να την εκφράζουν και δεν θα πρέπει να τιμωρούνται από τον νόμο. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Μπαρό για να τελειώσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. χώρα που γνωρίζω καλύτερα έχει ζήσει ε, έντονες αντιπαλότητες για αυτό το θέμα. Και προσωπικά θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει στα πλαίσια της ανεκτικότητας ε, και πράγματι και της ε, κατανόησης. Υπάρχουν οικογένειες που θέλουν να συνεχίσουν να διατηρούν τις ε, χριστιανικές τους παραδόσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βασιστεί στη συνύπαρξη των διαφορών. Συνεπώς νομίζω ότι έχουμε επενδύσει προβολικό χρόνο και προσπάθεια σε αυτό το θέμα. Στη χώρα μου εγώ έχω δει ότι και από τις δύο πλευρές επιδεικνύεται πολλές φορές ακρότητα ε, το θέμα όμω είναι ότι η συζήτηση αυτή δεν θα πρέπει να συμβαίνει εδώ. Θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα στην Γενική Συνέλευση Συμβουλίου τη Ευρώπη και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Όχι εδώ. Νομίζω ότι εκεί είναι η θέση αυτής της συζήτησης. Και εκ μέρους Κομισιόν ε, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι ασφαλώς η Κομισιόν είναι προσιλωμένη στην ε, προστασία της αρχής της σκεπτικής ελευθερίας και ασφαλώς θα δράσουμε ε, οποτεδήποτε υπάρχει περίπτωση ε, διακριτικής μεταχείρισης με βάση το θρησκεύμα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το νομικό πλαίσιο το οποίο μας επιβάλλουν οι συνθήκες. Η Κομισιόν δεν μπορεί να παρέμβει ως θεματοφύλακας των συνθήκων για θέματα τα οποία αφορούν ένα κράτος μέλος όταν αυτά τα θέματα δεν συνδέονται με το κοινοτικό δίκαιο. είμαι πολύ ειλικρινής. Η Κομισιόν σημειώνει τις αποφάσεις που ακούστηκαν, τις λαμβάνει υπόψη, αλλά δεν είναι δυνατόν να παρέμβει σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι σχετικό με το κοινοτικό δίκαιο. Το θέμα άπτεται της εσωτερικής ένωμης τάξης των κρατών μελών. Το λέω μία ακόμα φορά. Είναι χρήσιμη συζήτηση, είναι ενδιαφέρουσα παρόλο ότι πραγματικά θα ήθελα να ενθαρρύνω τους πρωταγωνιστές αυτής της συζήτησης να τηρήσουν το μέτρο. Ίσως το, η Γενική Συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης ε, θα μπορούσε με τη σειρά της να συζητήσει με έναν τρόπο πραγματικά πιο ωφέλιμο τι ερμηνείε που μπορούμε να δώσουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, όμω ε, εμεί, η Κομισιόν, ω θεματοφύλακα των συνθήκων δεν μπορεί να παρέμβει σε μια συζήτηση η οποία αφορά κατ' ουσίαν το Συμβούλιο τη Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να σα δώσω μια καλύτερη απάντηση σήμερα το βράδυ. Πρέπει όμω να είμαι ειλικρινή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. είναι θέματα τα οποία έχουν εμπίπτουν στην ένωμη τάξη του κάθε κράτους μέλους. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κλείνουμε έτσι τη συζήτηση. Και η επόμενη σύνοδος θα γίνει αύριο, θα λάβει χώρα αύριο από τις 9 ως τις 1 και από τις 3 ε, ως τις 7.